εβδομάδες από σήμερα στην Ολομέλεια των Βρυξελών. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο το πρωί στις 20 ε, Απριλίου Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 και από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις ε, 8 και μισή και από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα πρακτικά θα δημοσιευτούν και μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διαδίκτυο. Πέρα στις συνεδρίαση είναι 11 η ώρα. Καλό σας βράδυ, καλή νύχτα. <laughs>